everybody. We will continue uh, our uh, agenda with point 15. Σημείο 15 θα είναι το σημείο με το οποίο θα συνεχίσουμε τη μέση διάταξη. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Schengen 1 συν στο σύστημα Schengen 2. Ο εισηγητής μας είναι ο Κάλλος Κουέλιου. Θα του δώσω το λόγο για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσής του. Μετά θα ακούσουμε την άποψη της Κομισιόν και αν η Κυπριακή Προεδρία θέλει να πει κάτι. Βεβαίως, θα την ακούσουμε. Και μετά θα, θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κύριε Κουέλιου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη διεξαγάγει μια συζήτηση και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη να υπάρξει μια κοινοτική, μια ενωσιακή λύση και αρνείται τη συνέχιση του Σέγγιν κάτω από διακυβερνητική διακυβέρνηση. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο το Κοινοβούλιο πάντα υποστήριξε το ΣΥΣ 2. Η πρωτοβουλία που συζητούμε σήμερα κάνει, αποσαφηνίζει το νομικό πλαίσιο που έχει να κάνει με τη μετάβαση από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2 και επιτρέπει επίσης το νομικό πλαίσιο του ΣΥΣ 2 να εφαρμοστεί από τη στιγμή που το πρώτο κράτος μέλος θα εφαρμόσει την μεταφορά από το πρώτο σύστημα, τη μετάβαση από το σύστημα ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε νομική ασφάλεια και εμποδίζουμε προβλήματα να ανακύψουν στα κράτη-μέλη. Είναι επίση θετική η δυνατότητα ενωσιακής συγχρηματοδότησης δαπανών που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπομισθούν κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο. Είναι γεγονός ότι η καθυστέρηση με την οποία η Κομισιόν έχει παρουσιάσει αυτή την πρωτοβουλία δυσκολεύει τα κράτη-μέλη στο να καταφέρουν να εκμεταλλευτούν τη γραμμή του προπολογισμού η οποία προβλέπεται για τη μετάβαση αυτή από το ένα σύστημα στο άλλο και υποχρεώνται να εργαστούν σε ένα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο όπως και εγώ ο ίδιος που θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τη βοήθεια που μου παρέσχε στο έργο αυτό. Δυστυχώς στην τελευταία συναντηρία της Επιτροπής μας, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό δηλαδή, ε, τόνισα την λύπη μου γιατί το Κοινοβούλιο έτυχε απλώ αίτηση γνωμοδότησης δεδομένη τη πολιτική σημασία του θέματος αυτού και τη σημασία του και για τον προπολογισμό. Παρουσίασα παρόλα αυτά την πρόταση εκθεσής μου σε αυτή τη συνεδρίαση. Πέραν ορισμένων τώρα τεχνικών αλλαγών που μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητε. υπάρχουν και κάποιε αλλαγέ που έχω επιφέρει στην έκθεση μου καταρχήν σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, ώστε να υπάρξει ενίσχυση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική εποπτεία της πολύπλοκης αυτής διαδικασίας που είναι η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο να υπάρχει μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των τωρινών και των μελλοντικών αρχών που θα είναι αρμόδιες για την προστασία και την εποπτεία των δεδομένων ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Επιπλέον είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των δεδομένων αυτών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια στο SIS2. Τα προσωπικά δεδομένα φυσικά επέχουν μια ιδιαίτερη, περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και επομένω χρειάζεται να υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τη διαχείρισή τους ώστε να μην καταλήξει κάποιος να κατηγορηθεί αδίκως ή ακόμα και να κρατηθεί αδίκως μέσα στο χώρο του Σέγγεν. Το να διατηρήσουμε την ε, ακρίβεια και την αξιοπιστία των ε, στοιχείων που θα μεταφερθούν από το ένα σύστημα στο άλλο, αυτό είναι απαραίτητο και πρέπει να ληφθεί απαραίτητη μέρημνα. Πρέπει να γίνει επίση σαφέ ότι οποιαδήποτε στοιχεία ΣΥΣ 1 που δεν θα περάσουν στο ΣΥΣ 1 θα πρέπει να ε, καταστραφούν πλήρως μετά την περίοδο μετάβασης ώστε να μην παραμένουν αμφιβολίες ή νομικά κενά που να επιτρέπει να υπάρξουν ακόμα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην πρώτη φάση του ΣΥΣ και να παραμένουν εκεί μετά τη μετάβαση. Το ΣΥΣ 2 είναι ένα ουσιώδες εργαλείο για να ενισχυθεί η ασφάλεια του χώρου Σέγγεν για να σταματήσει η διακυβερνητική φάση του συστήματος του Σέγγεν και να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι το συς θα πρέπει να δει σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό και γι' αυτό το λόγο ζητώ την κατανόησή σας για το σφιχτό χρονοδιάγραμμα που είμαι υποχρεωμένος να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ. Πριν, πριν δώσω το λόγο σε αυτούς που ενδιαφέρονται, ίσως η Κομισιόν και η Προεδρία να θέλουν να λάβουν το λόγο. Κύριος Τουντοράς από την Κομισιόν. Uh, thank you very much, Mr. Chair. I'll try to be very brief. Uh, first of all, to acknowledge Ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα. Ε, πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο, ο οποίος έχει ε, κάνει πολύ σημαντική δουλειά για αυτή την έκθεση και εκ μέρου τη Επιτροπή θα τον ευχαριστήσω για την επικαδηματική του προσέγγιση ε, κατά την έναρξη των εργασιών επί αυτού του φακέλου. Δεύτερον, να ευχαριστήσω την ίδια την Επιτροπή που κατάλαβε το κατεπήγον της πρότασης και γιατί ήταν τόσο ε, κρίσιμη σημασία στο να περάσει όσο τον τον πιο γρήγορα για να έχουμε την καλύτερη δυνατή βάση για την μεταφάση από το ΣΥΣ1 στο ΣΥΣ2 που θα ξεκινήσει μέσα σε δύο-τρει μήνε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε την, ε, νομική, την ασφάλεια δικαίου ε, για αυτήν την διαδικασία. Ευχαριστώ λοιπόν τόσο τον κύριο Γοέλιο όσο και την Επιτροπή για, τον, τον τρόπο που χειρίστηκαν αυτό το φάκελο. Τώρα, κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για την έκθεση, για κάποια ζητήματα που ανέφερε ο κ. Κοέλιο, πρώτα για την ποιότητα των δεδομένων. Πράγματι, Αυτά συνδέονται και ε, από τα όσα αναφέρθηκαν ε, από την Επιτροπή. Ε, για αυτό το θέμα είναι απολύτως απαραίτητο η διαδικασία της εκαθάρισης των δεδομένων να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο πριν από την μετάβαση για να διασφαλίσουμε ότι μόνο τα σωστά στοιχεία και δεδομένα θα μεταφερθούν στο δύο. 2 Από πλευράς μας εμείς έχουμε ε, τον μετατροπέα, ο οποίο έχει ε, αξιολογηθεί και ελεγχθεί του τελευταίου 15 μήνε, για να είμαστε σίγουροι ότι μόνο τα σωστά στοιχεία θα μεταβιβάζονται στο ΣΥΣ2. Τώρα για την προστασία δεδομένων και την διαδικασία ε, κατά την ε, μετάβαση, συμφωνούμε ε, με τα όσα προτείνονται στην έκθεση. Είναι περίπλοκη διαδικασία. Ε, αυτή την εποπτεία την μοιράζονται και το EPPS και οι εθνικές αρχές. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτελούν ε, το ρόλο τους, ο καθένας το δικό του. για τις τροπολογίες ό,τι αφορά την ε, υποβολή εκθέσεων και την παροχή πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της ε, διαδικασίας της μετάβασης. Είναι ένα ελάχιστο εγχείρημα διαφάνειας. Βεβαίω και το παίρνουμε στα σοβαρά και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβαση, η Επιτροπή ε, θα ε, ενημερώσει το Κοινοβούλιο όπως αρμόζει για τα αποτελέσματα της διαδικασίας, για την τελική ημερομηνία. Ο μόνος τρόπος που δεν έχουμε εισαγάγει την ημερομηνία στο κείμενο βεβαίως και δεν είναι επειδή φοβόμαστε να δεσμευτούμε για την ε, θέσει σε λειτουργία του συστήματο. Απλώ ε, έτσι αφήνουμε ένα περιθώριο ε, στα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν ε, τι συμβαίνει, την κατάσταση και στο διάστημα που προβλέπεται από το ίδιο το κείμενο να ορίσουν την ημερομηνία θέση σε λειτουργία του συστήματος. Καταλαβαίνω ότι για τον κύριο Κοέλο και την Επιτροπή είναι σημαντικό να ορίσουμε ημερομηνία το σημειώνουμε και θα δούμε πώς ε, θα εξελιχθεί η συζήτηση σε αυτό το τομέα στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες, είμαι στη διάθεσή σας. Ερωτήσεις. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η Προεδρία ε, αναγνωρίζει το έργο του κυρίου Κοέλιο και της Επιτροπής ε, και θα προσπαθήσει όσο μπορεί να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν αυτός ο φάκελος. You Λάτφορντ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ότι ο κ. Κοέλιο έχει εργαστεί πολύ σωστά. Ξέρουμε ότι τα προγράμματα τη Σέγγεν βρίσκονται σε καλά χέρια και συμφωνώ απολύτω και με το συμπέρασμα ε, του αιτιολογικού σημειώματο, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα κρίσιμη σημασία εγχείρημα και μέσο ε, για την ε, περιοχή Σέγγεν που βελτιώνει συστηματικά και σημαντικά την προστασία δεδομένων και γι' αυτό θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να επιταχύνουμε τη δικασία. Περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό και ελπίζουμε επιτέλους τον Ιανουάριο να αρχίσει να λειτουργεί. Ελπίζω η αξιολόγηση του νέου συστήματος να καταδείξει ότι άξιζε τους πόρους που δαπανίσαμε ε, και θα κρατήσει και στο μέλλον χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Κοέλιο ότι η νομική βάση ε, που παρέχεται για τη διαβούλευση μόνο που προβλέπει μάλλον μόνο διαβούλευση είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Δεν γίνεται να έχουμε μόνο διαβούλευση ε, για κάτι που όπως είπα και ο κύριος Κοέλιο έχει πολιτική σημασία, δημοσιονομικές προεκτάσεις αλλά και ε, προεκτάσεις ό,τι φορά την προστασία δεδομένων. Επομένως είναι ανεπαρκές ε, το να έχουμε μόνο διαβουλεύσεις. Ε, επανερχόμαστε στις, ε, στον παλιό κακό καιρό πρώτη συναπόφασης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριο Κοέλιο έχει λάβει υπόψη ε, σημεία του EPPS για στοιχεία όπως η ε, επαλήθευση των δεδομένων ε, για τις τροπολογίες συγκεκριμένα 7 και 11 αναφέρομαι. Ιδίω ε, την έμφαση που δίνει στο γεγονό ότι όλα τα δεδομένα που δεν ε, μεταφέρονται από το, σύστημα, από το ΣΥΣ1 στο ΣΥΣ2 πρέπει να διαγράφονται. Και στηρίζω τις ε, προτάσεις που έχει κάνει για την ποιότητα των δεδομένων όπως πολύ σωστά λέει, οι συνέπειε των σφαλμάτων σε αυτό το τομέα για τα πρόσωπα μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η πρόταση δεν είναι σαφή σε ό,τι αφορά την ε, διατήρηση των δεδομένων. Ε, μιλάμε για διατήρηση των δεδομένων για ένα έως τρία έτη, αλλά για τα κράτη-μέλη δίνεται δυνατότητα ε, παράταση αυτού του χρονικού διαστήματος για όριστο χρονικό διάστημα για τις διαδικασίες παρακολούθησης που ε, τρέχουν ήδη. Τι ακριβώς καλύπτει αυτή η έννοια. Ορίζεται αυτό επαρκώς για να έχουμε αυτή την ασφάλεια δικαίου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας ε, πει δύο λόγια από αυτού ο εισηγητής. Ε, Γενικώ δεν υποβα... προτίθεμαι να υποβάλω τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρόταση, απλώς το επισημαίνω. Τέλος, ε, οι συνάδελφοί μου ξέρουν στην Επιτροπή ότι πάντα προσπαθώ να κρατήσω τη χώρα μου μέσα στα πράγματα, όσο αυτό είναι δυνατόν. Και ο εισηγητής πάντα ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα μιλήσω στην την Ιρλανδία βεβαίω, αλλά εν πάση περιπτώσει, Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ε, δικαίωμα opt-in. για αυτά τα δεδομένα, αλλά υπάρχει δυσκολία σε τη βάση. Από ό,τι κατάλαβα στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Κορεπέρ ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει δεύτερη ξεχωριστή πρόταση για τις ε, χώρες εκτός Σέγγεν που θα ε, προσχωρήσουν για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αυτή της πρότασης για να δούμε αν μπορεί και το Κοινοβούλιο να αντιδράσει με την ίδια ταχύτητα. Με έχουν διαβεβαιώσει ότι ο διαχωρισμός των δύο μέτρων δεν πρόκειται να καθυστερήσει ε, την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο δεύτερο σύστημα. Ελπίζω να μπορέσει να επιβεβαιώσει αυτή μου την εντύπωση και η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σάντσιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για την έκθεσή του. Να τον ευχαριστήσω επίσης γιατί μέσω των τροπολογιών που έχουν προταθεί έχει αρχίσει να θίγει τα πιο σημαντικά προβλήματα, την προστασία των δεδομένων, τον ρόλο τον οποίο θα πρέπει να έχουν οι εθνικές υπηρεσίες, οι εθνικές αρχές, συγγνώμη κτλ. Ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μία ημερομηνία ε, για να περνούν τα δεδομένα από το 6.1 στο 6.2. Έτσι θα δώσουμε την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη να έχουν μια συμπληρωματική δυνατότητα έτσι ώστε να ολοκληρώσουν την δημιουργία του, το πέρασμα των δεδομένων. Συμφωνώ επίσης και με την ανάγκη τακτοποίησης και καθάρισης πριν περάσουμε στην κατηγορία 6-2. Και όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο, Η datelor va putea fi menținută, mai ε, δεν έχουμε εγγυήσεις σχετικά με το κατά πόσον θα διατηρηθεί η ακαιρεότητα των δεδομένων και κατά πόσον πράγματι θα προστατευθούν τα δεδομένα αυτά. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί λάθος και δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να τα σβήσουμε ή όχι, αν τα διαγράψουμε ή όχι. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάποιες ε, αρχές, κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα είναι υπεύθυνε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή στην πρόταση ε, συμμετέχουν όλοι όσοι πράγματι μπορούν να συμμετάσχουν, μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα, εδώ θα τεθεί βέβαια και το θέμα της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας, γιατί είναι οι δύο χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο, δεν αναφέρονται. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ερμηνεύσουμε την 355 του 2010 και τη συνθήκη ένταξης των χωρών αυτών. Το καθεστώς αυτό λοιπόν της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας χρήζει διευκρινήσεων. Ο κύριος Πίρκλ είναι σαν μια ατέλειωτη ιστορία. Ένα σύριαλ. Έχει ξεκινήσει ήδη το 2006 η δημιουργία του Schengen 2, του ΣΥΣ 2, για να χρησιμοποιήσει την προσθέμενη αξία του Schengen, αλλά έχει κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κουέλιο, ο οποίος ε, ίσκησε την απαραίτητη πίεση για να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα αυτό και μπορούμε τώρα να ελπίσουμε ότι το 2013 θα λάβει πράγματι χώρα η μετάβαση των στοιχείων. Αυτό ελπίζω τουλάχιστον, μέχρι τότε όμως παραμένουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να διαλευκανθούν και εγώ πιστεύω αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Κουέλιο θέλω να το υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές για τα στοιχεία τα οποία θα μεταγραφούν και αυτό το οποίο έχουμε τονίσει στο παρελθόν για να αποφύγουμε μια σωρία προβλημάτων με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι ήδη λοιπόν απαραίτητο να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές για τα δεδομένα και να υπάρξει κάποια εκαθάριση των δεδομένων ώστε από το 2013 και επέκεινα να μπορούν να είναι αξιόπιστα τα σημεία αυτά. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία μετάβασης να τύχει της κατάλληλης εποπτείας και παρακολούθησης ώστε να γίνει σωστά η μεταγραφή των στοιχείων στο νέο ε, σύστημα και τα παλιά στοιχεία να εκαθαριστούν και να μην μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν. Εγώ έχω σκεπτικισμό γιατί αν αφήσουμε στα κράτη-μέλη την ε, ε, ευθύνη της μετάβασης μπορούν να προκύψουν προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρξει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την μετάβαση, το οποίο να είναι οριστικό, <clears throat> το κάθε κράτο να έχει δεσμευτεί μέχρι πότε θα πρέπει να κάνει τη μεταφορά αυτή στοιχείων από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2, ώστε το σύστημα 2 να μπορέσει να δημιουργήσει την απαραίτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να γίνει αποδεκτό ως ευρωπαϊκό εργαλείο ασφάλειας και ελέγχου. Είναι σαφείς λοιπόν οι προτάσεις που έχουν τεθεί, αλλά και εδώ αναφέρομαι προς την Κομισιόν περισσότερο και η ότι Κομισιόν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στα θέματα αυτά. Θα πρέπει η Κομισιόν να αναλάβει μια μορφή συντονισμού ώστε τα κράτη με ελεγχόμενο τρόπο θα μπορέσουν μέχρι την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος να δώσουν τα στοιχεία τους και τότε πράγματι θα είναι δικαιολογημένο να πούμε ότι υπάρχει ένα happy end μέσα στο 2013 σε αυτό το μακρύ σύριαλ. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Είναι μια ιστορία που μας απασχολεί πολύ καιρό το Σέγγεν ε, είναι πιο καυτά τα θέματα των συνόρων και πολλές φορές αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη έννοια κατεπήγοντος, αλλά είναι πιο αργές οι εξελίξεις σε σχέση με το σύστημα SIS2. Εμείς έχουμε τονίσει ότι είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει το σύστημα αυτό να είναι αξιόπιστο, αλλά θα πρέπει να τηρήσει και τις προδιαγραφές για τα, την προστασία των δεδομένων. Εμένα μου με έχει ευχαριστήσει ιδιαίτερα το γεγονό ότι ο κύριο Κουέλιο έχει υπογραμμίσει και πάλι την ανάγκη και τη σημασία τη προστασία των δεδομένων. Αλλά βλέπω ότι θα υπάρξουν προβλήματα με την μετάβαση από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2 θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρω και να γίνει σαφέ ποιες είναι οι πληροφορίε οι οποίες θα μεταφερθούν. Χρειαζόμαστε πράγματι όλε τι πληροφορίε που υπάρχουν στο ΣΥΣ 1 αν είναι κάποια στοιχεία τα οποία ουσιαστικά είναι πεπαλαιωμένα ή δεν είναι πια έγκυρα. Όλα αυτά συνδέονται με κάποια διαδικασία αξιολόγησης η δεν ειναι πια εγκυρα ολα αυτα συνδεονται με καποια διαδικασια αξιολογηση η οποια θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αποφύγουμε να μεταφέρουμε λανθασμένε πληροφορίε και θα πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα των αρμοδίων αρχών. Ποιοι θα αναλάβουν αυτό το έργο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε υπάρχει πολύ περιθώριο για αυθαίρετε ενέργειε στα κράτη-μέλη. Ο επόπτης ε, προσωπικών δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αν δούμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εμπλακούν με το σωστό τρόπο και τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση είναι να παραμείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο διαβούλευση. Αυτό είναι λανθασμένο. Γιατί και εδώ είναι ένα θέμα όπου δημιουργούνται ανάγκε για τον προπολογισμό Πρέπει επομένως να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται και με τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα ειδικό βάρος και όχι απλώς να την χάνει διαβούλευση από το Συμβούλιο για ένα θέμα το οποίο πια θα εντάσσεται στο ενωσιακό δίκαιο. Η κυρία Ντανόκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουν ακουστεί τα πάντα από τους συναδέλφους και τους συναδέλφους της δικής μου πολιτικής ομάδας. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κοέγιο για μια εξαιρετική προσπάθεια. Εμείς θα στηρίξουμε τις τροπολογίες που αφορούν την προστασία των δεδομένων την διαγραφή των δεδομένων, τη διάρκεια παρακράτησής τους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς αυτό. Ταυτόχρονα, σχετικά με την αποκατάσταση των προθεσμιών, στην 6 άρθρο 21, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, γιατί μέχρι τώρα παρά τις υποσχέσεις της Επιτροπής οι διαδικασίες δεν ήταν οι σωστές. Έχουμε το πρόβλημα το οποίο τίθεται in this dossier, but maybe you, you are more proficient in this and can answer. Για τη Βουλγαρία και τη Ρωμανία. Thank you. As there were questions to the Commission, I give back the floor to the Commission and then back to the Rapporteur. Υπήρχαν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της ξαναδίνω το λόγο και μετά το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε γιατί φέρατε στην επιφάνεια κάποια σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν σχετικά με το τι προτείνει το συγκεκριμένο έγγραφο και με το ποια είναι τα θέματα τα οποία προσπαθεί να λύσει. Καταρχάς, περίοδος κατακράτησης. Η περίοδος αυτή η οποία περιγράφεται στο 15 είναι αυτή που βασίζεται στην νομική βάση και η περίοδος παρακολούθησης βασίζεται στην νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Παρακολούθηση και έλεγχος σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος για τα δεδομένα συνολικά αλλά και τη λειτουργία του συστήματος. για την περίπτωση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου να απαντήσει στο θέμα, γιατί η πρωτοβουλία προέρχεται από αυτούς. Έχουν τεθεί και αρκετά θέματα σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων και με τα επίπεδα αποδοχής και τα κριτήρια μεταφοράς των δεδομένων στην κατηγορία 6.2. Δύο θέματα να διευκρινίσω εδώ. Κατάρχά η ευθύνη τη καταχώρηση των δεδομένων παραμένει στα κράτη-μέλη. Δεν έχει αλλάξει κάτι με το S2. Αυτό το οποίο προσπαθεί το νέο νομικό πλαίσιο να προσφέρει σε επίπεδο προστιθέμενης αξία είναι ότι η πρόσβαση στη νομική βάση είναι σε αυτή την περίπτωση κάτι που υπακούει σε ξεκάθαρους κανόνες σε σχέση με τον τρόπο καταχώρησης των δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων ή ενημέρωσή του και πιθανών αλλαγών. Λοιπόν, εδώ η προσφυγή λοιπόν και η χρήση ε, της νομικής βάσης θα είναι πιο εύκολη και θα συνεχίσει να υπάρχει. Ταυτόχρονα έχουμε συνεργαστεί με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών uh, σχετικά με την εφαρμογή των νέων επιπέδων ποιότητας ανταλλαγής πληροφοριών και από τις υπηρεσίες ΕΡΗΝ. Στόχος είναι τα δεδομένα, μόνο τα δεδομένα που σέβονται τους κανόνες της νομικής βάσης να εντάσσονται στο σύστημα και να υπάρχουν ε, κατά συνέπεια προσπάθειες ενημέρωσης ή διαγραφή σύμφωνα με τους κανόνες. Τώρα, για το τι δεδομένα μεταφέρονται από το ένα σύστημα στο άλλο. Οι νομικές βάσεις είναι αυτές για που μας λέγουν τι θα γίνει, το SAS2, θα συμπεριλάβει τα δεδομένα που προέρχονται από το 1, από το σύστημα 1 και ο μετατροπέας ο οποίος θα μετα... μεσολαβεί ανάμεσα στα συστήματα ακολουθεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες και διαγράφει τα δεδομένα που δεν ανταποκρίνονται στα προδιαγραμμένα ε, κριτήρια. Όλα λοιπόν τα δεδομένα θα περάσουν, αλλά τα δεδομένα τα οποία δεν θα ανταποκρίνονται στο φορμά, στη μορφή που έχει συμφωνηθεί, ε, θα τα μπλοκάρει ο μετατροπέας, ο ενδιάμεσος λογισμικός μηχανισμός. Οι πρωτοβουλίες θα ληφθούν πριν και κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου μεταβίβασης ε, νομίζω θα δώσουν εγγυήσει σε σχέση με την ακεραιότητα της διαδικασίας αυτής για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Τέθηκε από δύο από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι έχω απαντήσει εδώ στα πλαίσια της πρώτης συζήτηση που είχαμε λίγες εβδομάδες πριν. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία προς το παρόν δεν συμμετέχουν στο Σέγγεν δεν θα πάρουν μέρος στη διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων, έχουν πάρει μέρος σε όλες τις δοκιμαστικές λειτουργίες του SS2, τεχνικά είναι σε θέση δηλαδή να είναι μέρος, αλλά πλήρη συμμετοχή στο σύστημα θα γίνει μόνο τη στιγμή κατά την οποία ενταχθούν επίσημα στο Σέγγεν. Κάτι το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται πάντα σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο. Τώρα το Συμβούλιο θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Όχι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρους της ε, Προεδρίας ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να πω δύο λόγια. Πράγματι, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου πρότεινε το διαχωρισμό τη ε, πρόταση ε, για να διορθώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιρλανδία ε, στην μετάβαση στο καινούργιο σύστημα. Αυτό ο διαχωρισμό δεν έγινε για να αλλάξει κάτι επί τη ουσία τη πρόταση, αλλά για να αλλάξει η μορφή τη πρόταση. Όπως είπα, για να διευκρινιστεί καλύτερα η συμμετοχή των ε, δύο αυτών ε, κρατών μελών. Για το κατά πόσο τώρα αυτή η... αυτός ο διαχωρισμός της πρότασης ε, θα ενέχει και νέο γύρο διαβουλεύσεων στο Κοινοβούλιο. Όταν έγινε αυτός ο διαχωρισμός εξετάσαμε αυτό το ζήτημα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική τροποποίηση της ίδιας της πρότασης, απλώς τυπική ε, τροποποίηση για διευκρίνηση της συμμετοχής αυτών των δύο κρατομελών δεν απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση με το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπει και το δικαστήριο. Κατανοούμε ότι είναι σημαντικό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι θα ήθελε να δει και τα δύο μέσα μετά τον διαχωρισμό, παρόλο που δεν υπάρχει ουσιαστική τροποποίηση. Ε, ουσιαστικά έχουμε αντιγράψει, καταλέξει, ε, διευκρινίζοντας απλώς την, ε, το διαφορετικό καθεστώς συμμετοχής των δύο χωρών. Το Συμβούλιο προτίθεται να στείλει επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις ε, δύο νομικές πράξεις μετά το διαχωρισμό της πρότασης για να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να εξετάσει για τα δύο μέσα και να τα λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της τελικής νομοδότησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοέλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με υποστήριξαν και για τα θερμά λόγια που απίφθηναν σε μένα προσωπικά και θέλω να απαντήσω σε τρία θέματα, σε τρία ερωτήματα. Πρώτα, στο ερώτημα του κύριου Πίρκελ, λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε για την εφαρμογή του ΣΥΣ2. Γι' αυτό το λόγο στην εκθεσή μου εγώ προτείνω να υπάρξει ένας μήνας ως η προθεσμία για να γίνει η μετάβαση σε όλα τα κρατημέλη από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2. Το να αφήσουμε ένα ανοιχτό χρονικό πλαίσιο ή να αφήσουμε να πλανάται μια αμφισημία δεν θα επετύχανε τους στόχους ούτε της ταχύτητας ούτε της αποτελεσματικότητας. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ΣΥΣ 2 θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό. Ένα δεύτερο θέμα για το ερώτημα του κυρίου Ένσιου. Να πω ότι από τη δική μου πλευρά εγώ είμαι απόλυτα διαθέσιμος για αιτιολογικές σχέσεις οι οποίες θα εκφράσουν την ανησυχία όλων μας για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και είμαι στη θέση των για να βρούμε μια ικανοποιητική διατύπωση. Τέλος. Για αυτά που ανέφερε η Βαρονέσα Λότφορντ, και για τα οποία έδωσε μια απάντηση στο Συμβούλιο. Θέλω να πω το εξή, κυρία Πρόεδρε. Εμεί επισήμω δεν ξέρουμε τίποτα για την απόφαση του Συμβουλίου να κάνει το διαχωρισμό της απόφασης ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Από το State Watch το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε όμως επίσημα από τον Συμβούλιο είναι θλιβερό και πάλι ότι το Συμβούλιο δεν σέβεται το Κοινοβούλιο όπως θα έπρεπε όχι μόνο για λόγους καλής ανατροφής αλλά και για λόγους των ίδιων των συνθηκών. Όταν το Κοινοβούλιο μαθαίνει τις προθέσεις του Συμβουλίου με άλλους, από άλλες πηγές, τότε σίγουρα παραβιάζεται το πνεύμα των συνθήκων. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αν θα γίνει διαχωρισμός όπως λέει το State Watch ή όπως αναφέρεται στο σημείο 37 κάποια τροποποίηση. Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορηθεί για το θέμα αυτό πλήρως, εναπόκειται στο Κοινοβούλιο μέσα τη, μέσω της νομικής του υπηρεσίας να εξετάσει αν αυτή η ερμηνεία είναι έγκυρη ή όχι η ερμηνεία του Συμβουλίου. Εγώ δεν θέλω τώρα να προκαταλάβω αυτά τα θέματα προτού πάρουμε την επίσημη κοινοποίηση από το Συμβούλιο. Δεν θέλω λοιπόν από τώρα αν όταν πάρουμε αυτά τα στοιχεία τότε θα πρέπει να αποφανθεί η νομική υπηρεσία αν είναι απαραίτητη ή όχι η εκ νέου διαβούλευση του Κοινοβουλίου μετά από το splitting, το διαχωρισμό αυτό. Αλλά το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι το πρώτο όργανο το οποίο πρέπει να καταλάβει. Γιατί πρόκειται για πρόσβαση στα κράτη-μέλη ταμείων τα οποία θα καλύψουν το κόστος της μετάβασης, θα πρέπει να κατανοήσει το Συμβουλίο ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτά τα κονδύλια, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υποστήριξη όλων των συναδέλφων που θέλω να ευχαριστήσω και ιδίω τον εισηγητών. Αν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να επιταχύνει τη διαδικασία, δεν θέλουμε να υπάρχουν άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία είναι τα κατά κύριο λόγο εμπλεκόμενα, τα οποία θα θέσουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη νομοθετική διαδικασία και να εγκρίνουμε την πρόταση όπως μας έχει επισήμως παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ κύριε Κουέλιο, είναι σαφές αυτό που είχατε να πείτε προθεσμία για τις τροπολογίες. Τώρα σε αυτή την έκθεση είναι 24 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι και στις 11 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 16, στην μέση διάταξη, η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειες της στην αγορά εργασίας, η εξωτερική διάσταση του συνδεσμού, της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Φίλιπ Κλάις είναι ο εισηγητής. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έχει προετοιμάσει μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας είναι συνδεόμενη Επιτροπή βάσει του άρθρου 50 στην γνωμοδότηση αυτή και σήμερα θα, θα υπάρξει μια σύντομη παρουσίαση από τον, την εκπρόσωπο της Κομισιόν για την ενσωμάτωση ηθαγενών τρίτων χωρών και θα ακούσουμε και την άποψη του εισηγητού του κυρίου Κλέισ και θα ακολουθήσει συζήτηση. Δίνω το λόγο καταρχήν στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, first of all, I would like to thank you for taking up the issue of integration. Σας ευχαριστούμε που θέσατε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί τα θέματα αυτά συζητιούνται πολύ συχνά στο Συμβούλιο και καλό θα είναι να γίνει μια τέτοια συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η ενσωμάτωση, η ένταξη αν θέλετε, αυτό που προέρχονται από τρίτες χώρες είναι μια μακρά διαδικασία η οποία γίνεται σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στις πολιτικές ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης βοηθώντας την κοινωνική συνοχή και βοηθώντας έτσι και την ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τη νέα νομική βάση την οποία θέτει η συνθήκη της Λισαβόνας που αποκλείει μεν από τη μία την εναρμόνιση, από την άλλη βοηθά την ενίσχυση μέσων που λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν παρουσιάσαμε το 11 την σειρά προγραμμάτων για την ενσωμάτωση και ένταξη των μεταναστών τις συνθήκες ε, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως οι ε, εκπρόσωποι, οι πολίτες από τρίτες χώρες μαθαίνοντας τις γλώσσες και νιώθοντας ότι ανήκουν και αυτοί στις συγκεκριμένες κοινωνίες. Προβλέπουμε ας την ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων των μεταναστών. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης και για την επικύρωση ακριβώς των γλωσσικών ικανοτήτων, την αύξηση της συμμετοχής επίσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Επ' αυτών των βάσεων λοιπόν θα πρέπει και οι μετανάστες να συνεισφέρουν έτσι θετικά και στη δημιουργία του δικού τους μέλλοντος αλλά και της νέας χώρας που τους φιλοξενού. και σε επίπεδο τοπικής δράσης λοιπόν προτείνουμε μέτρα. Στην ουσία αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό εκ των κάτω προς τα άνω, συνεργαζόμενοι με την Επιτροπή των Περιφερειών. Κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως είπαμε, οι πολιτικές αυτές ενσωμάτωσης είναι πολιτικές που ανήκουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και έχουν τα μέσα για να το κάνουν. Μπορεί λοιπόν η κοινοτική νομοθεσία να δώσει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο όχι μόνο για τις συνθήκες εισόδου και παραμονής αλλά και σε σχέση με τις δυνατότητες ενσωμάτωσης, ένταξης και να υπάρξουν κοινοί κανόνες γιατί την από κοινού και ισότιμη αντιμετώπιση των μεταναστών. Το θέμα της άδεια εργασίας, σαν παράδειγμα, έχει συζητηθεί τα θέματα των δικαιωμάτων των εποχιακών εργαζομένων κτλ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και άλλους τομείς δράσης στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των πολιτικών ενσωμάτωσης, ανταλλαγής γνώσεων και χρηματοδότησης. Προτείνουμε επίσης να εμπίνουμε και στην εμπλοκή των χωρών προέλευσης για την διευκόλυνση της ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης των μεταναστών. Η ενσωμάτωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί βέβαια να ξεκινήσει από τη χώρα προέλευσης, αλλά κάποια μέτρα πριν την αναχώρηση μπορεί να βοηθήσουν ενημερώνοντας τους μετανάστες για το πώς να έρθουν στην Ένωση, ενημερώνοντάς τους για τις θεωρήσεις και παίρνοντας πληροφορίες και για τις χώρες τις οποίες θα πάνε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει επίσης το πλαίσιο για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης ανάπτυξης δικτών για τον έλεγχο της πολιτικής αυτής. Έχουμε αντιμετωπίσει τέσσερις τομείς, απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνικός αποκλεισμός, η καταπολέμησή του και συμμετοχή στα πολιτικά θέματα και στα κοινωνικά θέματα. Βλέπουμε ας πούμε ότι το ποσοστό των μεταναστών είναι κατά 10% συνήθως μεγαλύτερο από το ποσοστό των εργαζομένων γενικότερα στην Ένωση και αυτό είναι κάτι το οποίο συναντάμε και σε άλλους δείκτες τους οποίους χρησιμοποιούμε. Στο παρελθόν προετοιμάσαμε εγχειρίδια προς χρήση των εταίρων οι οποίοι συμμετέχουν στη διαχείριση των διαδικασιών ένταξης. Αυτή τη στιγμή εμείς δημιουργούμε τα λεγόμενα πεδία αναφοράς σε τρεις τομείς. Πρώτον τομέας γλωσσικών ικανοτήτων, δεύτερον υποδοχή από την τοπική κοινωνία και τρίτον συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής δραστηριότητας. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενσωμάτωσης με 25 δις ευρώ. Ήδη λειτουργήσε από το 2007 μέχρι το 2013. 60 προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από την κοινότητα και μέσω των εθνικών προγραμμάτων εμείς θα πρέπει να τονίσουμε και το προτείνουμε αυτό την τοπική διάσταση των μελλοντικών ρυθμίσεων για τη χορήγηση ασύλου. Να μην ξεχνάμε επίσης και την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των μεταναστών και τις πολιτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ένταξης των μεταναστών η συνεργασία με την Οικονομική και ε, Κοινωνική Επιτροπή ε, διοργανώνουμε δις τον χρόνο ένα φόρουμ ενσωμάτωσης και συμμετέχουμε στο φόρουμ αυτό φυσικά. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 16 και 17 Οκτωβρίου και θα έχει ε, τον τίτλο «Συμμετοχή των μεταναστών στη νέα οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» οι δυνατότητες τις οποίες δίδουν τα 22.500.000 μετανάστες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σήμερα στην Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σμιτ. Ο κύριος Κλάης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ανέβαλε να συντάξει μια τέτοια ε, γνωμοδότηση. Ως ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφασίσαμε να κάνουμε μια τέτοια γνωμοδότηση. Αμέσω μετά υπήρξε συνεδρίαση μεταξύ των γραμματιών και των δύο επιτροπών ε, για να προσδιορίσουμε ποια στοιχεία πρέπει να τα αναλάβει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και ποια η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία αποτελούν ζητήματα ευμερισμένης αρμοδιότητας και των δύο επιτροπών, ε, όπως η ε, νομοθεσία κατά των διακρίσεων, ενωσιακή πολιτική μετανάστευση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι οι κοινωνικο επιπτώσεις ε, της μετανάστευσης, η ένταξη των μεταναστών ε, στην ε, αγορά εργασίας, καταπολέμηση της φτώχειας, και οι δικέ μα αρμοδιότητε είναι τα δικαιώματα των μεταναστών, οι γενικέ πτυχέ τη ένταξη των μεταναστών και των ετούντων άσυλο, τα δικαιώματα, το καθεστώς και οι υποχρεώσεις των μεταναστών και ο συντονισμός των κρατών μελών ε, για την ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών. Βεβαίω πρέπει να ε, έχουμε κατά νου όσο γίνεται περισσότερο αυτόν τον ε, προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων, αλλά πράγματι το πρόβλημα με την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι τόσο ευρύ που είναι δύσκολο να το εντάξουμε στις αρμοδιότητες της μιας ή της άλλης επιτροπής. Για να μπορέσουμε να ασχίσουμε μια πολιτική ε, μετανάστευσης ε, με δημοκρατικό χαρακτήρα και νομιμοποίηση στη συνείδηση του πληθυσμού, πρέπει να εστιαστούμε όχι μόνο στα δικαιώματα, αλλά και ε, στις υποχρεώσεις. Θα επανέλθω σε αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο σε ένα ε, ε δικαίου που λειτουργεί σωστά, είναι σημαντικό η φυστάμενη νομοθεσία να εφαρμόζεται. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω ότι θα έχουμε μόνο αυτή την έκθεση για τους νόμιμους και όχι για τους παράνομους μετανάστες. Επίσης, για την ε, ανεξέλεγκτη εισρωή μεταναστών σε κάποια κράτη-μέλη, θα ήθελα να αφαιρθώ, που πλέον ε, απειλεί και την ικανότητα απορρόφησης αυτών των κρατών μελών για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ε, ή να υποδεχθούν αυτούς τους μετανάστες αλλά και να τους εντάξουν στην αγορά εργασίας. Υπάρχει λοιπόν και ανεξέλεγκτη μετανάστευση Υπάρχει βέβαια το θέμα της ε, επανένωσης των οικογενειών. Πολλές φορές ε, μέσω γάμων προσπαθούν να έρθουν ε, στα κρατημέλη μας και φαίνεται τελικά πολύ συχνά ότι δεν είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι άνθρωποι να, να ζήσουν σε μια ξένη χώρα και καταλήγουν στο σύστημα, στο κράτος πρόνοιας και δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε μέσα στην έκθεση. Η Επιτροπή απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων στη δική της ε, έκθεση, η οποία δεν είναι διαθέσιμη προ το παρόν, θα βασιστεί λοιπόν σε μεγάλο βαθμό αυτή η έκθεση σε μια μελέτη που έχει αναθέσει αυτή η Επιτροπή για την ένταξη των μεταναστών και τον αντίκτυπο της ε, ε, στην αγορά εργασίας και εκεί θα καταφανεί ότι ε, δίνεται μεγάλη έμβαση στο πρόβλημα των διακρίσεων, ότι θα πρέπει να υπάρξει πιο αυστηρή εφαρμογή της ε, νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, που βέβαια δεν θα υπάρχει διαματηρία για κάτι τέτοιο, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε και κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Ε, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπου, έτσι ισχύει και για τους μετανάστες. Και πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί εύκολα λέμε ότι όλα τα προβλήματα με την ένταξη των αλοχθώνων και των μεταναστών στην ε, αγορά εργασίας είναι εύκολο να, τα, ε, να λέμε ότι είναι πρόβλημα διακρίσεων. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στο Βέλγιο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ε, ισχυρή και κατασταλτική μάλιστα νομοθεσία κατά των διακρίσεων ε, και πολύ επίοικης ε, πολιτική ό,τι αφορά την, το πρόβλημα της ένταξης ε, των μεταναστών. Δεν μιλάμε τόσο για υποχρεώσεις, μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για δικαιώματα. Και βλέπουμε λοιπόν σε μια τέτοια χώρα όπως το Βέλγιο ότι Ακριβώς ε, εκεί λοιπόν το πρόβλημα της ένταξης στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα οξύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες ε, χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το πρόβλημα είναι τόσο σημαντικό όσο στο Βέλγιο, ε, όπου τόσα παιδιά καταλείπουν το σχολείο. Πρέπει αυτό να συνδεθεί και με την πολιτική που ακολουθείτε και που ασκείτε μια τέτοια γενναιόδορη και επίοικης ε, πολιτική που τελικά έχει ε, το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Γιατί δεν ε, τονίζουμε αρκετά την προσωπική ευθύνη των μεταναστών. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα ακραίο παράδειγμα ότι μέχρι πρόσφατος στο Βέλγιο έπρεπε κάποιος να, έχει μία, να, γνωρίζει μία από τις δύο ε, γλώσσες, επίσημες γλώσσες του Βελγίου. Βεβαίως τώρα βλέπουμε και ποια είναι η πραγματικότητα που είναι ε, μάλλον διαφωτιστική ίσως και βεβαίως και δυσάρεστη και έτσι προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια στοιχεία αυτής της πολιτικής όπως ε, υλοποιείται και απευθύνω έκκληση προς τους αδέλφους να μην κάνουν τα ίδια λάθη όπως αυτά που έχουν γίνει στο Βέλγιο. Αυτά είναι τα κέρια σημεία που θα ήθελα να υπογραμμιστούν στην έκθεση. Βεβαίως και θα δούμε και ποια είναι η θέση της Επιτροπής για το τι πρέπει να εξετάσουμε στη συνέχεια και περιμένω και τις ε, αντιδράσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλέης. Να δώσουμε το λόγο πρώτα στην κυρία Χίρς που είναι υπεύθυνη ε, για αυτήν την ε, έκθεση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση βλέπονται και οι δύο επιτροπές ε, εξετάζουν το θέμα της μετανάστευσης γιατί είναι θεμελιώδους σημασία θέμα και αφορά πολλούς τομείς, ε, αγορά εργασίας και εκπαίδευση, πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτή η έκθεση θα είναι πολύ σημαντική για αυτή τη νομική πράξη και ελπίζω να ε, αποστείλουμε κάποια μηνύματα. Στη δική μου επιτροπή βεβαίως και επικεντρωνόμαστε τόσο περισσότερο στην ένταξη στην αγορά εργασίας και σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Και θέματα όπως αυτά, όπως και η, η έλλειψη εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται συνήθως από την πλευρά μιας πολιτικής ασφάλειας, αλλά κυρίως υπό την ε, οπτική γωνία της οικονομικής πολιτικής, της απασχόλησης και φυσικά και υπό το, το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας που κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολύ καιρό. Επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει αυτή η έρευνα σαν βάση για την έκθεση αυτή, αλλά υπάρχουν και ανακοινώσει της Κομισιόν που έχουν ένα ευρύ πεδίο που καλύπτουν. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την Κομισιόν για την εργασία και την υποστήριξη που έχει λάβει, έχει παρουσιάσει, αλλά είναι πράγματι πολύ πλοκό και πολύ σχηδές το θέμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών και πρέπει να ληφθεί υπόψη με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε όλοι τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι επίμαχα στα κράτη-μέλη από τη μία μεριά τις υποχρέωσεις των μεταναστών, από την άλλη μεριά τα δικαιώματα των ε, μεταναστών. Είναι σωστό να έχουμε προσπάθεια μιας σωστής νομοθετικής ρύθμισης στα θέματα αυτά, τα οποία πρέπει επίσης να την χάνουν και σωστής εφαρμογής αυτά τα νομοθετήματα. Επομένως, εγώ μπορώ να αναφέρω ότι κατανοώ αυτά που λέει ο εισηγητής, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξουν εφαρμογές αυτών των προτάσεων από τους μετανάστες, από την άλλη μεριά πρέπει και το κοινωνικό σύνολο να δείξει μια ανεκτικότητα και μια κατανόηση των μεταναστών, κάτι το οποίο όλο και περισσότερο χάνεται με την οικονομική κρίση. Πιστεύω επίση ότι αυτή η εκθέση πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία τα οποία ίσω είναι καινοτόμα και ενδεχομένω και επίμαχα, αλλά πιστεύω το θέμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών όπου θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μονάχα ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Στη δική μου έκθεση θα υπάρξει μια πρόταση για να υπάρξει ένα εθελοντικό στη ε, σύστημα μορίων για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη με διάφορε μορφέ, έχουν τέτοια συστήματα. Εγώ θα μπορούσα να φανταστώ να υπάρξει εθελοντική δημιουργία ενός ε, τέτοιου συστήματος στα κράτη-μέλη και μπορούμε με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουμε περισσότερο σε μία μορφή κοινού συντονισμού και να εξάρουμε περισσότερο και την ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να είναι πολύ πιο ελκυστικές για τους μετανάστες και λόγω γλώσσας κυρίως από την Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει όμως να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα η οποία καλωσορίζει τους ανθρώπους που έχονται στην Ήπειρό μας και τους δίνει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν. Επομένως το θέμα δεν είναι μονάχα η ενσωμάτωση αφηρημένα, αλλά το πώς παρουσιάζουμε σε κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τη δυνατότητα να έρθει και να εργαστεί. Αυτά λοιπόν είναι σημεία τα οποία πιστεύω πρέπει να ενσωματωθούν στην έκθεση αυτή. Κάποιο άλλο σημαντικό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η, η παραδοσιακή, αν θέλετε, η, η σε βάθος γενναίων μετανάστευση. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μια χώρα και μένουν εκεί. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με το πρόβλημα αυτών οι οποίοι έρχονται, εργάζονται και φεύγουν. Και εδώ τίθενται πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνική ασφάλιση, με μεταφορά δικαιωμάτων κτλ. Και αυτό λοιπόν το στοιχείο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω, γιατί και αυτό αναφέρθηκε, είναι η παράτυπη ή παράνομη μετανάστευση. Φυσικά είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αφορά διότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και ένα από τα ζητήματα λοιπόν που πρέπει να διεξέλθουμε είναι οι άνθρωποι είναι εδώ παράνομα μεν, αλλά έχουν κάποια θέση εργασία, η οποία φυσικά είναι μη νόμιμη, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν να κερδίσουν το ψωμί του και να προσφέρουν κάτι στον εργασιακό χώρο και ίσω θα πρέπει να βρούμε τρόπου να δώσουμε σε αυτού του ανθρώπου τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους. Ξέρουμε ότι προσφέρουν κάτι στις κοινωνίες μας αυτοί οι άνθρωποι και επομένως θα χάσουμε κάτι άμα τους διώξουμε. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα σημεία επιπλέον που θέλω να αναφέρω στην εκθεσή μου, όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η αντιμετώπιση των φοιτητών που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα μετά το τέλος των σπουδών τους να βρουν μια θέση εργασίας. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν είναι σημεία τα οποία θα πελάβει η εκθεσή μου. Απλώς ήθελα να σας παρουσιάσω όλα αυτά τα στοιχεία για να εμπλουτίσω τη συζήτηση. Ο κύριος Σκούρια. Συγκράτησε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία μόνο παρατήρηση. Έχω την εντύπωση ότι όταν αναφερόμαστε στα θέματα της ενσωμάτωσης αναφερόμαστε κυρίως στους νέους και δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας το θέμα της εκπαίδευσης των νέων μεταναστών. Το λέγω αυτό γιατί πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα. Βλέπουμε νέα παιδιά τα οποία φτάνουν στο τέλος των σπουδών τους και τα οποία για λόγους κακής ερμηνείας του όρου αλληλεγγύη φτάνουν στο τέλος των σπουδών τους χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά την γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν. Δεν γνωρίζουν καν τους κανόνες ε, και τους νόμους. Ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο δεν γνωρίζει τους κανόνες και τους νόμους και τη γλώσσα μιας χώρας στην οποία μένει δεν θα βρει εύκολα δουλειά. Αυτό είναι λογικό. Είναι κάτι το οποίο έχω ζήσει γιατί πριν γίνω ευρωβουλευτής ήμουνα πρόεδρος μιας μικιό Ιταλικής η οποία ασχολείται με θέματα που αφορούσαν τα σχολεία στην Ιταλία και μεταξύ των οποίων και αυτό. Πολλές φορές παιδιά λοιπόν, τα οποία είχαν την δυνατότητα και τη βούληση να ενσωματωθούν, δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα να ενσωματωθούν, επαναλαμβάνω, τη γνώση της γλώσσας κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο στα πλαίσια της έκθεσης την οποία θα διατυπώσουμε στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εφόσον θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική δυνατότητα ενασχόλησης και απασχόλησης μάλλον των μεταναστών. Δύο μιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Λάμπερτ και Κάσμαν. Τζέιν και Μάικλ να είστε πολύ σύντομοι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο ή τρία σημεία. Μιλάμε για την ενσωμάτωση και όχι την απορρόφηση. Δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί εδώ μπορεί να ακολουθηθούν δύο διαφορετικοί δρόμοι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δύο θέματα νομίζω ότι θα πρέπει να προσθεθούν στα πλαίσια της συζήτησης αυτής. Όταν αναφερόμεθα στα θέματα της συμμετοχής, ένα σημαντικό κομμάτι των προτάσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν στις διάφορες εκθέσεις, τέθηκαν τα θέματα και των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και υπάρχει και το θέμα της διαφοράς των φύλων. Όταν βλέπει τις παλαιότερες εκθέσεις βλέπει ότι ένα πολύ σημαντικό των μεταναστών είναι γυναίκες και δεν έρχονται μόνο ως σύζυγοι, κάτι το οποίο πολύ συχνά βέβαια τις αντιμετωπίζουμε, αλλά αυτοδύναμα με τα δικά τους ε, δικαιώματα, με τη δική τους δουλειά και τα δικά τους ε, χαρακτηριστικά. Αυτό πολλές φορές ε, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας στη συζήτηση. Δεν αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες σαν ανεξάρτητους εταίρους και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Ιδιαίτερα σε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερ, το κύριο Κάσμαν. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Χαιρετίζω την πρόταση αυτή. Θέλω να πω επίσης ότι όταν εξετάζουμε τις κοινότητες των μεταναστών θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι μετανάστες από τους εργοδότες τους και από άλλους. Είναι ένα αμφίδρομο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά επειδή έρχομαι και εγώ από μια οικογένεια μεταναστών, η οικογένειά μου πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από πολλά χρόνια και ήμασταν κάθε άλλο παρακαλόδεκτοι εκεί θα πρέπει να πω για την τεράστια συμβολή των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης, τόσο στην πολιτική, κοινωνική, αλλά και οικονομική ζωή των χωρών μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μάικλ. Ερχόμαστε στο... Δεν θέλει ο εισηγητής να πει κάτι. Ε, εντάξει, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Το επόμενο σημείο είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 5ης Σεπτεμβρίου 5 Σεπτεμβρίου και λάβαμε αυτή την απόφαση σε σχέση με την ε, παρακολούθηση και την υποπτία των εξωτερικών συνόρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αντιταχθεί στο κείμενο αυτό, αλλά δεν είχε την κατάλληλη πλειοψηφία για να σταματήσει αυτό το μέτρο, αλλά η Επιτροπή μας ε, προσέφυγε στο δικαστήριο κατά του μέτρου αυτού, γιατί ξεπερνάει την εμβέλεια των μέτρων επιτροπολογία και αφορά και την ουσία των αποφάσεων που είχαν εγκριθεί σε, σε διαδικασία συναπόφασης. Ο Γενικός Αγγελέας έκανε την πρότασή του και ακολουθήθηκε στην τελική απόφαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2012 και θεωρεί ότι εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη δεν ισχύει η απόφαση αυτή μέχρι ότου εγκριθεί η επόμενη απόφαση. Δίνω το λόγο στην κυρία Ντίν τώρα να παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτής της απόφασης και θα ζητήσω μετά από την Κομισιόν να μας πει πώς θέλουν να αντιδράσουν σε αυτή την απόφαση του δικαστήριου και μετά θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για περαιτέρω συζήτηση. Κυρία Ντίν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, παρουσίασή σας. Δεν θα κάνω την εισαγωγή που ήθελα να κάνω και θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Το δικαστήριο έπρεπε να αποφανθεί επί δύο θεμάτων. Το ένα ήταν το θέμα του παραδεκτού σε διαδικαστικό επίπεδο και αυτό προκύπτει από το γεγονό ότι στην Ολομέλεια μια πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου ψήφισαν κατά του σχεδίου απόφαση, αλλά δεν επετέφθη η απόλυτη πλειοψηφία η οποία μπορούσε να αναστείλει την απόφαση αυτή. Και το μέτρο λοιπόν αυτό έγινε δεκτό. Το Συμβούλιο είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι εφόσον το δικαστήριο θα μπορούσε να είχε σταματήσει την απόφαση αυτή επί τη βάση του ότι ξεπερνούσε τις εξουσίες που προκύπτουν από τον κώδικα για τα σύνορα του Σέγγεν, δεν μπορεί τώρα το Κοινοβούλιο να επανέλθει και να καταθέσει μια προσφυγή για τα θέματα αυτά. Αλλά όπω και ο Γενικό Εισαγγελέας, το δικαστήριο θεώρησε ότι ήταν παραδεκτή αυτή η προσφυγή. Υπάρχει το δικαίωμα δράση του Κοινοβουλίου, το οποίο δεν μπορεί να εξαρτηθεί από μια απόδειξη του ενδιαφέροντου ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, ούτε επί τη βάση της τάσης που ανέλαβε όταν έγινε δεκτό αυτό το μέτρο. Το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην έγκριση αυτή τη απόφαση δεν περιορίζει και δεν αποκλείει τα δικαιώματά του να καταθέσει προσφυγή για τα θέματα αυτά. Επομένω, το δικαίωμα του δημοκρατικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να ανατραπεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένω, θεωρήθηκε διαδικαστικά παραδεκτή η προσφυγή. Το δεύτερο θέμα που έπρεπε να εξασφαλίσει το δικάστιο είναι αν αυτή η απόφαση θα μπορούσε νομίμως να εγκριθεί επί τη βάση του, των ε, εκτελεστικών εξουσιών βάσει του κώδικα του Σέγγεν. Αυτέ αυτές οι εξουσίες, οι εφαρμοστικές εξουσίες επιτρέπουν την έγκριση πρόσθετων μέσων σε σχέση με την εποπτεία. Αλλά βάσει του κώδικα μόνο ε, στοιχεία μη ουσιώδη μπορούν να εγκριθούν βάσει των εκτελεστικών εξουσιών. Το Κοινοβούλιο επιχειρηματολόγησε ότι αυτά τα στοιχεία ήταν πράγματι κέρια και ουσιαστικά και έπρεπε να εγκριθούν με συναπόφαση. Και το, και το δικαστήριο συμφωνεί με τη θέση του Κοινοβουλίου. Πρώτο, θεωρεί ότι οι ρήτρε και πρόνοιε οι οποίε αποτελούν πολιτικέ επιλογέ, οι οποίε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των νομοθετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να τύχουν εγχώρηση. Η αξιολόγηση του τι είναι ουσιώδε και του τι δεν είναι ε, ουσιώδε δεν μπορεί να τύχει εκχώρηση, ούτε παραμένει στην αποκλειστική δυνατότητα εκτίμησης της νομοθετικής εξουσίας. Θα πρέπει να βασίζεται αντίθετα σε παράγοντες αντικειμενικού χαρακτήρα που να μπορούν να τύχουν νομικού ελέγχου. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ο χαρακτήρας και οι ιδιαιτερότητες του τομέα στον οποίο αναφερόμαστε. Εξήτασε μετά το δικαστήριο το έβρος εφαρμογή και, το και το νόημα του άρθρου 12 του κώδικα Schengen και σημείωσε το άρθρο 12 του κώδικα ευρεία τη ενία ε, ζητά από τις αρχές να εμποδίσουν τις ε, παράνομε διελεύσει των συνόρων, να αντιμετωπίσουν τη διαμεθοριακή εγκληματικότητα και να πάρει μέτρα εναντίον ατόμων που έχουν περάσει παράνομα τα σύνορα. Αλλά το άρθρο 12 με αφηρημένο μοναχα τρόπο περιλαμβάνει τα καθήκοντα των σύνοροφυλάκων και δεν έχει καθόλου κανόνε σε σχέση με τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία οι συνοροφύλακε έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν εναντίον ατόμων ή εναντίον ε, πλοίων όταν συλλαμβάνονται. Αντίθετα, το παράτημα της ε, απόφασης αυτής θεσπίζει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να αναλάβουν οι συνοριοφύλακε εναντίον πλοίων τα οποία ε, διακριβώνονται και των ατόμων που επιβαίνουν. Μπορούν τα πλοία να σταματηθούν, να υπάρξει επιβίβασή τους και να υπάρξει και έρευνα και κατάσχεσή τους. Η απόφαση επίσης αυτή δίνει και τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις για την έρευνα και την διάσωση πλοίων και ατόμων που βρίσκονται στα πλοία αυτά. Το δικαστήριο θεώρησε ότι η απόδοση τέτοιων εξουσιών στους συνοριοφύλακες έχει σαν αποτέλεσμα πολιτικές επιλογές οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των νομοθετικών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι επιλογές σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει σωστή στάθμιση των αντιμαχόμενων συμφερόντων και επομένως με τον τρόπο αυτό μονάχα μπορούν να αποδοθούν εξουσίες στους συνοριοφύλακες και τις συνθήκες χρήσης των εξουσιών τους. Επιπλέον και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των εμπλεκομένων ατόμων μπορεί να παραβιαστούν σε σημαντικό επίπεδο Εάν μπορεί να γίνει αυτό σε σημαντικό επίπεδο, μάλλον συγγνώμη, τότε θα πρέπει να επιληφθούν οι νομοθετικέ εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το Συμβούλιο συμφωνεί με το Γενικό Εισαγγελέα και θεωρεί ότι η απόφαση αυτή περιλάμβανε ουσιαστικά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να εγκριθούν παρά μόνο από την νομοθετική εξουσία. Επίση, απέριψε την άποψη του Συμβουλίου ότι μη δεσμευτικέ κατευθυντέ γραμμέ δεν θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ουσιαστικά στοιχεία. Γιατί αυτέ οι γραμμέ ήταν τμήμα του λειτουργικού σχεδίου των επιχειρήσεων τη Frontex και έπρεπε να υπάρξει μόρφωση με αυτέ. Επομένω, απέρριψε την απόφαση αυτή και την ακύρωσε στο Συμβούλιο, αλλά διατηρεί τα αποτελέσματα αυτή τη απόφαση, όπω ζήτησε το Κοινοβούλιο, μέχρι ότου σε ένα λογικό επίπεδο μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή ε, ρυθμίσει οι οποίε θα αντικαταστήσουν αυτή την επίμαχη απόφαση. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια νέα νομοθετική πρόταση από την Κομισιόν και οι νέοι κανόνε θα πρέπει να εφαρμοστούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ω συνομοθέτε. Η απόφαση του Συμβουλίου επίση δίνει κατάλληλη κατεύθυνση για τη χρήση του άρθρου 290 τη Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι κατεξουσιοδότηση πράξη και εκεί που χρησιμοποιείται και η ιδέα, η αρχή των μη ουσιδών στοιχείων. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τα ερωτήματά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει πώς σκοπεύουν να δράσουν μετά από την απόφαση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, δεν έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση αυτής της σημαντικής απόφασης η οποία κυκλοφόρησε, δημοσιεύτηκε μάλλον εδώ και δύο εβδομάδες. Πρέπει να παρατηρήσουμε καταρχάς ότι το δικαστήριο ακολούθησε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την συνέχιση της ισχύω της απόφασης και δεν έχουμε πλέον προβλήματα νομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα υπάρχουν και αρκετά θέματα που πρέπει να αναλυθούν ιδιαίτερα με το, σχετικά με το πώς θα ε, ε, ερμηνευτεί το θέμα της εμβέλειας και τι αυτό σημαίνει για το μέλλον. Και τρίτον, είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι η απόφαση αυτή καλύπτει ορισμένα πάρα πολύ περίπλοκα θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν ή δεν μπορούν να ληφθούν στα διεθνή ύδατα κτλ και στόχοι της απόφασης αυτής ήταν σημαντικοί και εξακολουθούν να είναι, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Frontex, να υπάρχει επίσης νομική διαφάνεια για τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυση μας την οποία θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν και είμαστε διαθέσιμοι και εδώ για να ακούσουμε τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων μεταξύ των οποίων και της δικής σας επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Yes, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τις νομικές υπηρεσίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σε πρώτο στάδιο πολύ ε, σωστές συμβουλές μας έδωσαν επί του θέματος, γιατί η νομική υπηρεσία μας έδωσε, ε, μας συμβούλευσε και βάσει αυτών των συμβουλών η Επιτροπή μας πήρε την πολιτική απόφαση να ε, προσφύγει στο δικαστήριο για αυτό το θέμα. Ε, με ανακούφιση ε, διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο δικαιώθηκε και η Επιτροπή μας δικαιώθηκε σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της απόφασης της Συμβουλίου που τώρα έχει ακυρωθεί. Βεβαίως ε, θα περίμενα περισσότερες πληροφορίες για το τι προτίθεται να κάνει τώρα η Επιτροπή. Έχουμε απόφαση Συμβουλίου που έχει ανακληθεί. Παρόλο που διατηρούνται οι νομικές ε, διαστάσεις της παρόλο, μέχρι την αντικατάστασή της. Ποια όμως είναι η πολιτική θέση της Επιτροπής, ε, πώς προτίθεται να αλλάξει αυτή την απόφαση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Επιτροπή για την υποβολή μιας ε, κατάλληλης ε, πρότασης που βεβαίως θα βασίζεται στην, ε, στην απόφαση αυτή τη φορά. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή να είναι λίγο πιο ακριβής και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει σήμερα, να μας πει πότε προβλέπετε να είναι σε θέση να μας δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Κάσμαν που ήταν εισηγητής ε, επί του ζητήματος. Ε, τότε. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως δεν ε, συμμερίζομαι αυτή την εφορία, αν μπορώ να πω, του συναδέλφου. Γιατί αν είχαμε ακολουθήσει τις διαθέσεις του Κοινοβουλίου του 2010 το Μάρτιο, δεν θα είχε τεθεί σε ισχύ ε, αυτή η, απόφαση και δεν θα είχαν διασωθεί τόσοι άνθρωποι τόσο αποτελεσματικά ε, τόσοι άνθρωποι είχαν πέσει στη θάλασσα, τόσο ναυαγοί ε, και όλα αυτά εξαιτία ε, των επιπτώσεων ε, αυτή τη απόφαση. Τότε, ω εισηγητή, αναγνώρισα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υπερβεί τι εξουσίε τη Πράγματι, το αποδέχθηκα και με τη συνάδελφα Μαγκιντίν, με την οποία συνεργάζομαι τόσα χρόνια. Αποδέχθηκα λοιπόν την απόφαση, την εγγνωμοδότηση της ε, νομική υπηρεσία, ότι δηλαδή το Συμβούλιο είχε ε, ακολουθήσει τη λανθασμένη νομική βάση, όμως και τότε το έλεγα και με, ε, με δικαίωσε και ο Γενικό Αγγελέα και η απόφαση ότι αυτές οι διατάξει είναι απαραίτητε, πρέπει να διατηρηθούν και δεν πρέπει να δίνουμε νομικέ ε, μάχε ε, σε βάρο μεταναστών που πνίγονται στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε να διατηρηθεί η απόφαση γιατί θεωρούμε ότι τα νομικά επιχειρήματα μπορούμε να τα λύσουμε στη συνέχεια και πολύ χαίρομαι. Με ικανοποίηση μπορώ να σα πω ότι έχουν λυθεί. Επίσης, με ικανοποίηση μπορώ να σα πω ότι οι ε, επιπτώσεις της απόφασης, ε, κατόπιν της απόφασης του δικαστηρίου, θα ε, μείνουν σε ισχύ μέχρι την θέση σε ισχύ νέων κανόνων και έτσι δίνουν στην Επιτροπή την πολυτέλεια του χρόνου να υποβάλει νέα μέτρα που θα τύχουν τις στήριξη του Κοινοβουλίου. Σίγουρα με τα ε, ε, θα αναγνωρίσουν συνάδελφοι το ε, σημείο 3 της απόφασης ότι θα πρέπει το Συμβούλιο να, τα έξοδα μάλλον να βαρύνουν το Συμβούλιο. Σίγουρα η ομάδα μου θεωρεί ότι έχει δικαιωθεί. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Χωρί να επαναλάβω τα όσα ε, υπόθηκαν προηγουμένω, έχω κάποια ερωτήματα ειδικότερα προ την Επιτροπή. Το θέμα του χρόνου είναι πολύ σημαντικό. Το δικαστήριο είπε ότι πρέπει να υποβληθεί νέα πρόταση ε, εντό ευλόγου χρονικού διαστήματο. Επομένω, ε, εγώ αυτό το ερώτημα θα σα κάνω. Πότε θα υποβληθεί η νέα πρόταση. Έχουν ήδη περάσει δύο εβδομάδε από την απόφαση του δικαστηρίου. Ε, σίγουρα δεν είναι αρκετό χρονικό διάστημα για να συντάξετε μια νέα πρόταση, αλλά μπορείτε να μας πείτε περίπου τι θα γίνει και πότε. Και ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε για τη νέα πρόταση από την παλιά πρόταση. Ε, επίσης, θα ήθελα να μου πει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για το ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι επιπτώσεις για την απόφαση Ε, και τι συμβαίνει με, τους, ε, με την απόφαση για τους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι ο λόγος στην Επιτροπή. Thank you. Well, I'm I can't... Ευχαριστώ. Ε, φοβάμαι δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι έγκυρα μένα, αλλά πολύ δύσκολα. Θα επανέλθουμε στην Επιτροπή μας το ταχύτερο δυνατό με ένα χρόνο διάγραμμα. Αλλά κατά δεύτερο λόγο, και εγώ κατανοώ αυτό το οποίο ελεγχθεί για την ανάγκη να δούμε τα διδάγματα από την εμπειρία της ε, εφαρμογής αυτής της απόφασης τα τελευταία 2,5 χρόνια και να συνδέσουμε καλύτερα αυτή την απόφαση με άλλα εργαλεία τα οποία είτε είναι υφιστάμενα είτε είναι στο στάδιο των προτάσεων δεν είναι εύκολο για μας μέσα σε δύο εβδομάδες να πούμε πώς θα έχει μια προτινόμενη νέα απόφαση. Και δεύτερον θα χρειαστούμε, όπω είπα προηγουμένω να ακούσουμε όλου του εμπλεκομένου και αυτό θα περιλαμβάνει φυσικά την Επιτροπή σα στη Λίβη αλλά και τα κράτη-μέλη, ίσω και την ίδια την υπηρεσία του Frontex για να δούμε ποια είναι τα διδάγματα τα δικά του. Τι πιστεύουν για την εφαρμογή των αποφάσεων μέχρι στιγμή, αν χρειάζεται να αλλάξουν αυτά ή όχι. Και αυτό θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Και θα επανέλθουμε όταν μπορούμε το ταχύτερο δυνατό με ένα γενικό πλαίσιο ε, για το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να ερμηνεύσει, αν είναι κάποιο νομομαθή που ξέρει τι σημαίνει λογικό, εύλογο χρονικό διάστημα, όπω λέει η απόφαση του δικαστηρίου, θα ήθελα να το ξέρω. Κυρία Κέλλερ, θέλετε να επανέλθετε. Αυτό ακριβώ είναι το ερώτημά μου προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ίσως τι ακριβώς είναι τα όρια του εύλογου χρονικού διαστήματος τι ακριβώς μπορεί να πει και η κυρία Ντίν για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Δεν έχω μια πρόχειρη απάντηση, αλλά υπάρχουν ε, περιπτώσεις, υπάρχει κάποια νομολογία και μπορώ να επανέλθω και να σας πω είναι, ποια είναι η νομολογία για τα θέματα αυτά, το ιστορικό του δικαστηρίου. Κύριε Κάσμαν δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει το Κοινοβούλιο από το να υιοθετήσει το δικό του χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πόσο επαρκής είναι ο χρόνος που χρειάζεται. Νομίζω όμως ότι η λογική του επομένου θέρους, όπου οι άνθρωποι πράγματι θα περάσουν σε παλιό... Και σαν πιο κάραγα, για να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό τίποτα δεν μας εμποδίζει να ζητάμε τακτική ενημέρωση. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Ψάχνουμε τον εισηγητή του επόμενου θέματος, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται, είναι εδώ και δεν θα υπάρξει διάλειμμα. Θα περιμένουμε να έρθει όμως. Και μετά έχουμε άλλα δύο θέματα. Ευχαριστώ Μόνικα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση γιατί έχουμε εδώ μια έκθεση με 459 κατατεθειμένες τροπολογίες. Λυπάμαι για τη Μόνικα που είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει και όλες αυτές τις τροπολογίες. Το θέμα λοιπόν είναι η εξέταση των ε, τροπολογιών που έχουν ε, κατατεθεί στην έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, περίοδος 10 ε, με 12 και όπως είπα οι τροπολογίες είναι πραγματικά πολλές. Ευχαριστώ. Θα ομιλήσω την Σλοβακική, λέει η κυρία Μπένοβα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. για αυτή την πάρα πολύ σημαντική για τις σημαντικές αστροπολογίες που καλύπτουν πάρα πολλά θέματα και θα πρέπει ακριβώς γι' αυτό το λόγο να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμά μας, κάτι το οποίο θα επιτρέψει όχι μόνο σε μας, αλλά στο σύνολο του Κοινοβουλίου να προετοιμαστεί σωστά για την ψηφοφορία. Πριν ξεκινήσω τα σχόλιά μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην προηγούμενη Ολομέλεια, ο Πίτροπος Βέντλινγκ πρότεινε κάτι, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και η έκθεσή μου άλλωστε το λέει, όπως και οι δικές σας τροπολογίες. Τι είναι αυτό η αξιολόγηση των δικαστικών συστημάτων, των συστημάτων δικαιοσύνης που ισχύουν σε όλες τις χώρες. Έχω εδώ τον λεγόμενο πίνακα επιδόσεων δικαιοσύνης, το οποίο θα είναι αν θέλετε ουσιαστικά το σύμβολο της κατάστασης του κράτους δικαίου. Αύριο έχουμε με την κυρία Ρέντινγκ μία συνάντηση και νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να υποστηρίξουμε κάποιες συμβιβαστικές συμπληρωματικέ τροπολογίες γύρω από τον πίνακα επιδόσεων έτσι ώστε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να παίξει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της συγκεκριμένη διαδικασίας. Θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες αυτές. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες ε, συμπληρώνουν αν θέλετε αυτά τα οποία λέγω εγώ για τις ευρωπαϊκές αξίες και για την ανάγκη προστασίας τους. Σε επίπεδο γενικών συστάσεων έχουμε λάβει πάρα πολλές προτάσεις με τροπολογίες οι οποίες κάνουν και πρακτικές προτάσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μέσω ακριβώς των μελετών επιπτώσεων που γίνονται για την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και σχετικά πάντα με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να παίξουν ένα σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των δεδομένων. Το θέμα είναι λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι συμβατές με αυτές τις αξίες και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει βελτίωση της συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά όργανα που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, με τα εποπτικά μέσα που έχουν όλες οι χώρες και με τους διεθνείς οργανισμούς. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις εμπλέκουν και τον φορέα για την παρακολούθηση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και όλα αυτά πρέπει να να συμπεριληφθούν και στο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο αναφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες οι οποίες συνάπτονται επίσης και με το πρόβλημα των Ρωμά, με την αντιμετώπιση των διακρίσεων, με την προστασία των μειονοτήτων. Όλες αυτές οι προτάσεις λοιπόν εστιάζουν περισσότερο στις πιο κριτικές πτυχές αυτής της προβληματικής περιοχής και μπορώ να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο εμπλουτίζουν και την εκθεσή μου. Εμείς εργαζόμαστε επί τη βάση των τροπολογιών αυτών με στόχο να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές ε, οι οποίες θα αντανακλούν και τη συζήτηση στην Επιτροπή μας αλλά και τις πρώτερες αποφάσεις της ε, Ολομέλειας. Οι αποφάσεις ας πούμε για τους ε, Ρωμά ή οι αποφάσεις για μειονότητες κτλ. Πολλές ε, φορές πρόκειται για μειονότητες ή για μετανάστες. Πολλοί συνάδελφοι εκφράζουν και μία ματέωση όταν η διαδικασία αυτή βασίζεται σε μία έλλειψη ή δεν βασίζεται μάλλον σε επαρκή αλληλεγγύη. Είναι απαραίτητο για μας να δώσουμε και ε, την απαραίτητη έμφαση στο κεφάλαιο για την Ιθαγένεια και να εξασφαλίσουμε και τις προϋποθέσεις για να υπάρξει δυνατότητα εφαρμογής των ρητρών σε αυτό το κεφάλαιο. Επίσης η Επιτροπή μας θα πρέπει να εξασφαλίσει και πάλι τη συμμετοχή σας στην επανεπεξεργασία του πλαισίου για, την, για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες σε σχέση με, το, με τα κεφάλαια της πρότασης, αλλά υπάρχουν, πιστεύω, οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Αν ο στόχος μας είναι να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα είναι εφαρμόσιμα τα θετικά ε, στοιχεία της πρότασης αυτής και θα μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό τρόπο, τότε μπορούμε να έρθουμε σε συνεργασία με τους ε, σχεδόν εισηγητές και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε από κοινού να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συμβαστικές λύσεις οι οποίες θα συγκροτήσουν μια ισορροπημένη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάσμαν πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πριν υποσχέθηκα ότι θα είμαι σύντομο, τώρα θα είμαι ακόμα πιο σύντομο. Να ευχαριστήσω τη Μόνικα για την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει και για το συνεκτικό τρόπο με τον οποίο έχει εξετάσει το θέμα της εφαρμογής και τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως θα ήθελα να την ευχαριστήσω που τόνισε κάποιες ε, παρεξηγημένες μειονότητες όπως είναι οι ομοφιλόφιλοι και ούτω καθεξής. Από πολιτικής πλευράς μπορώ να πω ότι έχω ξαναβρει τον ύπνο μου. Ευχαριστώ. Εφόσον είμαι σκιώδης από πλευράς ΕΛΚ, θα ήθελα να πω ότι θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για το έργο σας. Όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρία, ήταν εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης και κατανοώ τη δυσκολία της, ε, του χειρισμού τόσων τροπολογιών. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι επικεντρώνονται σε ορισμένα ζητήματα. Υπάρχει δυνατότητα συμβιβαστικών τροπολογιών και τις περιμένουμε με ανεπομονησία. Και με ικανοποίηση βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσε τροπολογίε για τα δικαιώματα των ε, παιδιών ε, και τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε ε, καλούς συμβασμούς. Παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα. Ας συνεχίσουμε τώρα. Η κυρία Ντανόκα. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τη Μόνικα και από εσάς που δεν άκουσα την παρέμβασή σας γιατί καθυστέρησα. Άκουσα όμως τα όσα είπε η Α, την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Κα, κατά τη συνάντηση των ε, σχεδόν θα, ε, θα βρούμε και μια κοινή θέση για τις κοινέ τροπολογίες. Βεβαίω έχουμε διαφορετικέ απόψει ω πολιτικέ ομάδε, γι' αυτό υπάρχουν και τροπολογίε. Τώρα, για τις τροπολογίες ε, που κατέθεσα εκ μέρου της ομάδας των Βρασίνων, επαναλαμβάνουμε τη θέση που έχουμε περιγράψει και σε προηγούμενες εκθέσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε τέτοια εργαλεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, για την, για την περιφερειακή χάρτα γλωσσών. Για τη χάρτα περιφερειακών γλωσσών μάλλον Υπάρχουν περιορισμοί και επιφυλάξεις. Τότε θα πρέπει να αποσυρθούν μέχρι να τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις. Υπάρχει τροπολογία για την παράγραφο 17. Εγώ Υποβάλλω έκθεση αύριο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε αυτή την έκθεση πρέπει να τονίσουμε τον ιδρυτικό κανονισμό και την ανάγκη αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού ε, του Οργανισμού θεμελιών Δικαιωμάτων Ο βασικός στόχος είναι η διεύρυνση της εμβέλειας της εντολής αυτής. Η πρόταση της Επιτροπής να διευρύνει ε, την ε, εντολή ε, του Οργανισμού Θεμελιών Δικαιωμάτων ώστε να συμπεριλαμβάνει και την αστυνομική συνεργασία δεν έγινε ε, δεκτή ω πρόταση από το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο αναφέρθηκε και η πρόθεση να εξεταστεί και το θέμα των εθνωτικών μειονοτήτων, αλλά Δεν υπήρξε στήριξη, αλλά παραμένει η πρόθεση. Και εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να διαβρινθεί και όχι να περιοριστεί ε, η εντολή αυτού του οργανισμού θεμελιώδων δικαιωμάτων. Βεβαίως, εκρεμεί πρόβλημα σε τρία κράτη-μέλη για τους ε, απάτριδες. Εσθενία, Σλοβενία και Λιθουανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της διάλυσης του Ομοσπονδιακού κράτους. Και έχουμε πλέον ανθρώπους ε, ε, ε, υπό ειδικό καθεστώς που θεωρούνται απάτριδες και στη Λετωνία ε, πάνω από τους μισούς, στη Λιθουανία, όχι, στη Λετωνία, συγγνώμη, πάνω από τους μισούς έχουν γεννηθεί. Στη Λετωνία δεν έχουν όμως δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εκλογές. Ούτε να εκλεγούν στη δημόσια διοίκηση και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ αυτών των πολιτών και των ε, υπολείπων. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα ε, του, αν αυτοί θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, γιατί συνήθως καλύπτονται από τη λετωνική πρεσβεία. Αν όμως δεν υπάρχει λετωνική πρεσβεία, τότε τι συμβαίνει. Βεβαίως και πρέπει ε, αυτοί οι πολίτες όπως και οι υπόλοιποι λετωνοί πολίτες να έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν σε μια άλλη πρεσβεία. Όμως και πάλι έτσι δεν επιλύονται τα προβλήματα των απάτριδων. Και χαίρομαι που η συγγήτρια θίγει αυτό το ζήτημα στην έκθεσή της. Τη συγχαίρω λοιπόν και πάλι και της εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ξαναδίνω το λόγο στη Μόνικα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο. Θέλω και μια ακόμα φορά να τονίσω ότι η έκθεση αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και αύριο στην συζήτηση με την κυρία Ρέντινγκ. Εγώ είμαι έτοιμη να συζητήσω μαζί της αυτά τα θέματα και να θέσω ερωτήματα και θα είμαι πολύ ικανοποιημένη αν μπορεί να υπάρξει μια έκθεση που θα προέλθει από εμά που αφορά όλες τις θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπένοβα. Η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα λάβει χώρα στις 10 και 11 Οκτωβρίου στη συνεδρίασή μας. Και τώρα χρειάζεται ένα σύντομο διάλειμμα. Γιατί ούτε ο εισηγητής ούτε οι σκιώδεις εισηγητές για το επόμενο θέμα έχουν εμφανιστεί. και επομένως θα συνεχίσουμε στις 5.30 λέει η πρόεδρος. Για να περάσουμε στη συζήτηση του σημείου 19. Πρώτο Θεός στις 5.30 λοιπόν. Μετά από μια μικρή διακοπή, το επόμενο θέμα Έχουμε τον κύριο Μπουσουτήλ, εισηγητή για την έχει ζητηθεί να ξεκινήσουμε έκθεση πρωτοβουλίας γύρω από το θέμα αυτό και τις ρήτρες αλληλεγγύης. Αμοιβαία άμυνα, λοιπόν, ρήτρες αλληλεγγύης για αμοιβαία άμυνα, πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις. Λοιπόν, εισηγητής ο κύριος Μπουσούτηλ. Θα του δώσω το λόγο πρώτα. Και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους βουλευτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με το θέμα του χρονοδιαγράμματος αυτής της γνωμοδότησης. Είναι κάτι που έχει άμεση σχέση θα έλεγα για το αν θα έχουμε πραγματικά μια γνωμοδότηση στο τέλος ή όχι. Για να δώσουμε λοιπόν εγκαίρως τη γνωμοδότησή μας στην ΑΦΕΤ, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη, μία επιλογή έχουμε, να προχωρήσουμε με τη γνωμοδότηση αυτή το ταχύτερο δυνατόν, μόνο στα αγγλικά, μόνο στην αγγλική γλώσσα και να ψηφίσουμε ήδη στην επόμενη συνάντηση της ΛΥΜΠΕ στις 11 Οκτωβρίου. Γνωρίζω ότι αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους συναδέλφους, περιορισμούς ουσιαστικά, αλλά το χρονοδιάγραμμα της ΑΦΕΤ αυτό είναι. Και αν δεν εμείνουμε, δεν έχει κανένα νόημα να υπάρξει αυτή η γνωμοδότηση. Το θέμα είναι λοιπόν ή θα προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα και μόνο στην αγγλική ή δεν θα υπάρξει γνωμοδότηση. Πέραν τούτου, και δέχομαι βέβαια, παρακαλώ τους συναδέλφους να δεχθούν τους περιορισμούς αυτούς και περνάω στα θέματα ουσίας. Πρώτον, περί τίνος πρόκειται. Οι ρήτρες αλληλεγγύης, όπως γνωρίζουν είμαι βέβαιος οι συναδέλφοι, αναφέρονται στο άρθρο 222 της συνθήκης και εισάγουν νομικές υποχρεώσεις δεσμευτικές για κάθε κράτος μέλος να βοηθάει το ένα το άλλο στην περίπτωση που υπάρξουν μείζονες, μείζονος μορφής δυσκολίες όπως τρομοκρατικές ενέργειες και είτε φυσικές καταστροφές είτε ανθρωπογενείς καταστροφές. Αυτό το άρθρο της συνθήκης, το οποίο είναι νέο, πρόσφατο, καθιστά δυνατόν για πρώτη φορά για τα κράτη-μέλη να βοηθούν το ένα το άλλο. Και αυτή είναι υποχρεωτική αλληλεγγύη πρέπει να βοηθήσουν το ένα κράτος μέλος το άλλο έχουν τη νομική υποχρέωση πλέον μέσω της συνθήκης. Για να μπορέσει λοιπόν το συγκεκριμένο άρθρο αυτό να αποκτήσει ουσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια νομοθετική πρόταση για να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες αποφάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να συγκεντρώσω την προσοχή μου στα επόμενα σημεία και θα εκτιμούσα φυσικά παράλληλα τη συνεισφορά των συναδέλφων ήδη από τώρα και θα είμαι βέβαια σε επαφή και με τους σκιώδεις εισηγητές μετά από τη σημερινή παρουσίαση. Τα θέματα λοιπόν τα οποία εγώ περιλαμβάνω στην γνωμοδότηση είναι τα εξής. Πρώτον, συνδυασμός των προσπάθειών και πόρων από όλα τα κράτη-μέλη. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη σήμερα είναι υπεύθυνα για την διαχείριση των κρίσεων στο εδαφός τους. Όμως, οι καταστροφές πάρα πολλές φορές είναι διαμεθοριακού χαρακτήρα και επιβάλλουν συμμετοχή για την αντιμετώπιση τους άνω του ενός κράτους μέλους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκείς πόρους και μέσα έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν το άρθρο 222 καθιστά τον εφικτό τον συνδυασμό των δυνάμεων και των πόρων των διαφόρων χωρών. Δεύτερον, θέτω το θέμα του συντονισμού των διαθεσίμων ευρωπαϊκών μέσων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει θα έλεγα ε, μια μεγάλη καλή γκάμα μέσων που μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση αντιμετώπισης ε, τρομοκρατικών ε, υποθέσεων κτλ. Επιθέσεων, συγγνώμη, φυσικών καταστροφών, Europol, Frontex, Eurojust, όπως και η δύναμη ανταπόκρισης σε έκτακτες κρίσεις και καταστροφές. Όλα αυτά λοιπόν τα μέσα τα οποία υπάρχουν, όλες αυτές οι υπάρχουσες οντότητες θα πρέπει να συντονίζονται έτσι ώστε η εντολή την οποία λαμβάνουν να διεκπεραιώνεται σωστά και να μπορεί να βοηθήσει όταν χρησιμοποιείται και γίνεται αναφορά στην ρήτρα αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφύγουμε φυσικά και την επικάλυψη των διαθεσίμων μέσων και δεν θα πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικά μέσα τα οποία να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα ήθελα επίσης να προτείνω να αντιμετωπίσουμε το θέμα το πότε η ρήτρα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται. θα πρέπει άμεσα να χρησιμοποιείται η διαδικασία, να ξεκινάει η διαδικασία, θα πρέπει να ξεκινά όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες απόκρισης που έχει και τι σημαίνει αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα του πότε ο μηχανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Μόνο σε καταστάσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η δυνατότητα αυτή σε πολλαπλές περιπτώσεις, εφόσον πάντα μιλάμε για κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέσω αφορά το πόσο μπορεί η χρήση του άρθρου 222 να γίνεται προληπτικά και όχι απλά εκ των υστέρων. Η ιδέα μου είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με την απόκριση σε μια επίθεση, σε μια καταστροφή, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την βελτίωση της συνεργασίας έτσι ώστε να προλαμβάνονται τέτοιου είδους καταστάσεις και να μην συμβαίνουν. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν εδώ δυνατότητες σύνδεσης της ρήτρας αλληλεγγύης και μια σωστή στρατηγική για την αποτροπή των τρομοκρατικών ενεργειών σαν παράδειγμα. Τέλος, αλλά παραμένει κάτι το σημαντικό, στην περίπτωση θα μπορούσε το άρθρο αυτό να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί για κατεπίγουσες καταστάσεις που προκαλούνται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που μερικές φορές δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί βέβαια να θεωρηθούν καταστροφικές αλλά παρόλα αυτά δημιουργούν δευτερευόντως ουσιαστικές δυσκολίες για ορισμένες χώρες. Σαν παράδειγμα πέρυσι 50.000 άνθρωποι έφτασαν στην ίσο Λαμπεντούζα. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο γεγονός ε, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κανονικά. Λοιπόν, προσπάθησα να είμαι σύντομος, έκανα μια σύνθεση των θεμάτων τα οποία θα ήθελα να σας θέσω και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω τους συναδέλφους και να επανέλθω ίσως αργότερα κλείνοντας τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία με έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσφατα ανέλαβα το ρόλο της σκιώδης ηγητρίας για το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να σας πω την ευτυχία μου όταν πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα και θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδης εισηγητής. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα όπου υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και έλλειψη εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που οδηγούν στην κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη της αλληλεγγύης και η αλληλεγγύη πρέπει πράγματι να αποκτήσει την πλήρη σημασία του. Πολλά πράγματα υπάρχουν στη συνθήκη της Λισαβόνας και καλά και χρήσιμα. Αν μονάχα τα εφαρμόσαμε όπως έπρεπε. Τα άρθρα όπως η ρήτρα αμοιβαία αρρωγής και αλληλεγγύης δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτό είναι λυπηρό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό και προσβλέπω στις προσπάθειες που θα το αλλάξουν αυτόν. Υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείες που καλύτερα θα τους αντιμετωπίσουμε από κοινού, όπως είπε και ο εισηγητής, εθνικές, φυσικές καταστροφές σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρύτερο επίπεδο και είτε είναι ανθρωπογενείς είτε φυσικές οι καταστροφές, επειδή επηρεάζουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προς το συμφέρον μας να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ιδίως όταν ξεπερνούν τις ικανότητες ενός μοναχακράτους μέλους να τα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Πολλές φορές οι καταστροφές αυτές είναι διαμεθοριακές, θα έπρεπε να μπορούμε και να τις προλάβουμε όταν είναι αυτό δυνατό και να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τομεί σε πολλά κράτη-μέλη όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την αλληλεγγύη και με το να έχουμε ένα συστηματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας και να μεταλαμβαδέψουμε τις βέλτιστες πρακτικές μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Δεν είμαι εμπειρογνώμη για το θέμα αυτό. Μόλις ανέλαβα αυτά τα θέματα, αλλά προσβλέπω στη συνεργασία με τον κύριο Μπουσουτήρ για το θέμα αυτό και στη στενή συνεργασία με τους άλλους ηγητές και είναι χρήσιμο να δώσουμε και τις δικές μας θέσεις προς την Επιτροπή ΑΦΕΤ για την εφαρμογή της ρήτρα αλληλεγγύης. Αυτό είναι μια πρόκληση για την Επιτροπή μας και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα του κυρίου Μπούσουτιλ, να απαντήσω μάλλον στο θέμα του κυρίου Μπούσουτιλ, για μένα για, στο, στο βωμό της ταχύτητας είμαι έτοιμη να δεχτώ και τη χρήση μόνο των αγγλικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι με το θέμα αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν με πειράζουν τα αγγλικά εμένα. Είναι καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Χαιρετίζω αυτό που είπε ο κύριος Μπούσουτιλ. Νομίζω ότι θέτει πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ τώρα θέλω να τονίσω ότι οποιαδήποτε απάντηση θα πρέπει να έχει τον αναλογικό χαρακτήρα. Γιατί αυτό που είναι βασικό είναι να ξέρουμε ποια είναι η κλίμακα στην οποία θα λάβουν όλα αυτά τα γεγονότα. Τι είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνάει τις εθνικές ικανότητες και ποια είναι μια ανάλογη απάντηση. Και αυτό μας ενδιαφέρει όλους, είτε ασχολούμεθα με θέματα αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που θέλουμε μια αναλογική αντιμετώπιση, αλλά όχι μια αντιμετώπιση που μπορεί να οξύνει περισσότερα τα πράγματα. Πρέπει επίσης να υπάρχει σαφής λογοδοσία, αν θέλουμε, να υπάρξει συνεργασία διαφόρων φορέων και οργανώσεων. Θα πρέπει να είναι σαφές από τη δική μας πλευρά ποιος έχει την ευθύνη για την συνολική διαχείριση αυτών των καταστάσεων Έχουμε δει στο παρελθόν τι έχει γίνει σε σχέση με κινήσεις για την ε, αντιμετώπιση μεταναστευτικών ρευμάτων όπου δεν είναι σαφές ποιος ε, έχει την ε, αρμοδιότητα και δεν υπήρξε σαφής λογοδοσία και δεν ήταν σαφής ποιος ήταν υπόλογος σε ποιον. Το άρθρο για την ε, αλληλεγγύη μιλάει επίσης και για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών από μια τρομοκρατική επίθεση. Για μας θα ήταν ίσως χρήσιμο να είμαστε πιο επακριβείς σε σχέση με τη μορφή με την οποία θέλουμε να δούμε να υπάρχει αυτή η προστασία, με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την προστασία και να τη συνδέσουμε με πιθανές κυβερνοεπιθέσεις αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αρκετά ζουμερή έκθεση από την Επιτροπή μας μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα και μπορούμε να τονίσουμε ότι πράγματι υπάρχει πέρα από τη λογοδοσία και ένα θέμα δημοσίων ελευθεριών εφόσον συζητάμε για την αλληλεγγύη και τη ρήτρα αλληλεγγύης και κατανοώ ότι πολλές φορές στο παρελθόν δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική η έκφραση της αλληλεγγύης. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε σημαντικά τις ενεργειές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζέιν. Δεν ζητά κανείς άλλο τον λόγο. Επομένω, Σάιμον, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ήθελα μόνο να πω ότι τίποτα δεν με κάνει πιο περήφανο ως Ευρωπαίο πολίτη από το να βλέπω ε, την Ευρωπαϊκή Σημαία πάνω ε, σε κουτιά ανθρωπιστικών αποστολών, ε, σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές. Και νομίζω ότι αυτό το αισθάνονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι πολίτες δεν θέλουν μόνο να δείχνουν την αλληλεγγύη τους σε περίπτωση επιθέσεων και καταστροφών, όμως νιώθουν περήφανοι να βοηθούν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Είναι λοιπόν ε, ευθύνη δική μας ε, να προωθήσουμε αυτό το μέσο, γιατί αν έχουμε το κατάλληλο νομοθετικό, είναι το, το κατάλληλο νομοθετικό μέσο ε, για την πρακτική εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και για το θέμα του χρονοδιαγράμματος του, του φακέλου και νομίζω, από ό,τι κατάλαβα, θα προχωρήσουμε με την πρόταση που υπέβαλα, δηλαδή να συντάξουμε το κείμενο μόνο στα αγγλικά και να τεθεί και προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και να πάμε για τις ψηφοφορία στη Λίμπη στις 11 Οκτωβρίου. Ελπίζω ε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα να στείλω στους συναδέλφους το σχέδιο γνωμοδότησης και για, την, για τις τροπολογίες ήρθα σε επαφή και με τη γραμματεία. Ε, νομίζω ότι είναι καλύτερο να βάλουμε ως καταληκτική ημερομηνία την 3η Οκτωβρίου. Και έτσι έχουν αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα και συνάδελφοι για να ε, καταθέσουν τις τροπολογίες τους. Ε, εν τω μεταξύ, βεβαίως και θα είμαι σε άμεση επαφή με τους ε, σκιώδεις για να συζητήσω τη γνωμοδότηση πριν ακόμα την παρουσιάσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών μόνο στα αγγλικά στις 3 Οκτωβρίου και ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή Λίμπες στις 11 Οκτωβρίου. κάνουμε διάλειμμα πάλι τώρα. Τώρα για το επόμενο σημείο της μερικής διάταξης, μάλλον θα πρέπει να το περάσουμε. We have 10 uh, more minutes until 6 o'clock. 10 λεπτά μας μένουν μέχρι τις 6. Σήμερα είναι το απόγευμα των διαλυμάτων. Ας κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα λοιπόν, μέχρι να έρθει ο κύριος Πρίμπε για να μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις